Και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Δήλωση της Κομισιόν για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 8 Απριλίου 2014 σε σχέση με τη διατήρηση δεδομένων και θα ήθελα να ζητήσω, από την, να την κυρία Επίτροπο Μάστρομ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου που ελήφθη πριν από καμιά δυο μέρες η Κομισιόν ε, χαίρεται για την ε, διασάφηση της, του δικαστηρίου για την ε, ισχύ της οδηγίας για τη διατήρηση των δεδομένων. Η απόφαση ε, επιβεβαιώνει κάποια από, τις, από τα συμπεράσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την εφαρμογή της οδηγίας του 2011 και είχαμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά πριν από δύο χρόνια με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η οδηγία αυτή δεν ε, συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και θα πρέπει να έχει δώσει περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες. Άλλα θέματα τα οποία θέτει το δικαστήριο είναι η πρόσβαση στη χρήση από τις εθνικές αρχές, ο ορισμός του σοβαρού αδικήματος της αξιοπινής πράξης, ε, μέτρα ασφάλειας, ε, περίοδος διαφύλαξης και ο τόπος διατήρησης των δεδομένων και η ανάγκη διαφοροποίησης μεταξύ ατόμων και τη σχέση τους με ποινικά αδικήματα και την ε, προστασία των επαγγελματικών ε, απορρίτων. Στην έκθεση της Κομισιόν ε, σχολιάσαμε και κάποια από αυτά τα θέματα. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η διαφύλαξη των δεδομένων δεν πλήττει από μόνη της τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το δικαστήριο μιλάει για την ανάγκη να σεβαστούμε την αρχή της αναλογικότητας και να έχουμε αυστηρές προϋποθέσεις, ούτως ώστε να γίνει σεβαστή αναγνωρίζει ότι κάποια όρια στα θεμελιώδη δικαιώματα θα μπορούν να δικαιολογηθούν στο όνομα των θεμητών και πραγματικών δικαιωμάτων, ε, συμφερόντων συγγνώμη, που είναι κατά πολέμη σοβαρών αδικημάτων και τρομοκρατία. Εμεί έχουμε ξεκινήσει την ε, σκέψη και τον προβληματισμό για το αν χρειάζεται μια νέα νομοθετική πρόταση και αν φυσικά γίνει κάτι τέτοιο, η επόμενη Κομισιόν θα προωθήσει αυτή την πρόταση. Θα, λέει το δικαστήριο θα πρέπει να γίνει γρήγορη μεταρρύθμιση της οδηγίας και κυρίως ε, τι θα γίνει με το σχέδιο οδηγίες που αφορά τον τομέα των διοκτικών υπηρεσιών. Ο κύριος Βέμπερ έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδεικνύει ότι η Ευρώπη έχει προχωρήσει, έχει ενισχυθεί. Φυσικά η πολιτική μπορεί να αποφασίσει το Συμβουλίο των Υπουργών, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτό το οποίο ελέγχει τι αποφάσει. Αυτό είναι σωστό. Η νομοθετική εξουσία να βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο τη δικαστική εξουσία. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μα πρέπει να τύχουν προστασία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό η νομοθετική εξουσία. Αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και θα ήθελα το υπογραμμίσω ενώπιον όλων των συναδέλφων και τα εθνικά κοινοβούλια, τα εθνικά δικαστήρια, συγγνώμη, θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία αυτού του μηνύματο, όπω έκανε το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην Καλσούη. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να προασπίσει τι αρχέ τη χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα πρέπει εμεί ω κοινοβουλευτικοί να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτή τη συλλογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών δικαιωμάτων που αφορούν την προσωπική ζωή των ατόμων και που περιλαμβάνει εδρεωμένη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλε σημαντικέ ελευθερίε για τι οποίε τονίζω και πάλι ότι ω πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Παραμένει βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα μεγάλο πρόβλημα το ότι και η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την πίεση της τρομοκρατίας. Υπάρχει μια απειλή τρομοκρατία, ε, τρομοκρατίας η οποία δεν έχει εξαλειφθεί αλλά δυστυχώς παραμένει. Υπήρξαν πολλοί νεκροί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και μαζί με αυτούς καταστράφηκαν οικογένειες, χάθηκαν μοίρες ανθρώπινες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαραίτητη προστασία των ε, πολιτών. Γι' αυτό τονίζω από την πλευρά του ΕΛΚ ότι ο κίνδυνο τη τρομοκρατία δεν έχει παρέλθει. Εξακολουθεί να υπάρχει η τρομοκρατία όπω και στο παρελθόν. Χρησιμοποιεί όλε τι τεχνικέ δυνατότητε που έχει. Ξέρουμε ότι ήταν ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη στη Μαδρίτη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως λέει και η Ευρωπόλ και το γερμανικό Bundeskriminalamt το, υπηρεσία αντιμετώπισης εγκληματικότητας τονίζει ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες και απαραίτητες οι ε, πληροφορίες από τις συνδέσεις και η εκμετάλλευσή τους και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είπε ότι δεν πρέπει να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία πολιτών. Είπε όμως ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορεί να μειωθεί το μέγιστο διάστημα ε, διατήρησης αυτών των στοιχείων. Πρέπει να καταλήξουμε και σε κοινού ορισμούς σε σχέση με την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα. Να περιορίσουμε λοιπόν τη χρήση αυτών των στοιχείων για τα πιο σοβαρά εγκλήματα και να υπάρχει και η δυνατότητα των δικαστών να αποφασίσουν αν θα υπάρξει πρόσβαση ή όχι σε αυτά τα στοιχεία. Η τρέχουσα Κομισιόν θα είναι στην ε, θέση της μέχρι τον Οκτώβριο. Θα πρέπει λοιπόν να μην αναμειχθεί η Κομισιόν στην προεκλογική εκστατεία, αλλά να λάβει το καθήκον του να εκπονήσει μια νέα πρόταση και να θέσει τη νέα αυτή πρόταση ενώπιον του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μια νέα ρύθμιση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα νομικό κενό. Παραμένουν αυτή τη στιγμή οι εθνικές ρυθμίσεις ενισχύ και θα πρέπει να παραμείνουν για όλους αυτούς που θέλουν να προστατεύσουν τους πολίτες. Αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο για τη συλλογή και τη διατήρηση των ε, προσωπικών στοιχείων. Πρέπει όλες οι χώρες να υπακούν σε ένα κοινό σύστημα και όχι να έχει καθεμία το δικό του σύστημα γιατί αυτό δεν οδηγεί στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών θεμελιωδών ελευθεριών. Εμείς ως ΕΛΚ υποστηρίζουμε τα δικαιώματα αυτά, σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε και κατευθυντήρες γραμμές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που δεν θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Βέμπερ. Ο κύριο Μέρφη θέλει να σα ρωτήσει κάτι με μπλε κάρτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που... ευχαριστώ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Είπατε ότι η τρομοκρατία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Εγώ θέτω το ερώτημα κατά πόσο η τρομοκρατία είναι χρήσιμο εργαλείο για το Eurogroup, για την Επιτροπή, για όλους όσοι στην Ευρώπη θέλουν ε, να ε, υπονομεύσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, ε, το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα και απλώς χρησιμοποιούν την τρομοκρατία ως πρόσχημα. Δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση του επιχειρήματος αυτού της τρομοκρατίας. Αλλά δεν πρέπει και εσείς οι άλλοι συνάδελφοι από τη δική σας πτέρυγα να παραγνωρίζουν την ύπαρξη της τρομοκρατίας. Υπάρχει αυτή η απειλή και πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες. Είναι και τα δύο απαράγραπτα και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Η κυρία Εντφέλτ έχει το λόγο. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Μωράης πρώτα, για δυόμιση λεπτά. Δεν με πειράζει να με μπερδεύετε με την κυρία Νετφέλτ. Ίσως να πούμε και κάποια παρόμοια ε, πράγματα εκ μέρου ε, των σοσιαλιστών. Ε, δώστε μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω. Η οδηγία για την διατήρηση δεδομένων βεβαίω ιδρύθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπω ακούσαμε. Και από την ομάδα μα χαιρετίζουμε αυτή την ε, απόφαση. Βεβαίω ειδήθηκε εν μέσω δύσκολων συνθήκων, όμω είναι σημαντική και πέραν τούτου. Ε, Ποια άλλα ζητήματα υπήρχαν εκείνη την περίοδο που τώρα έχουν διορθωθεί και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και αυτό περάτηκε και η ομάδα μου. Η απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι οι φυστάμενοι κανόνες ε, δεν βρίσκουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μέτρων ασφαλείας και επιτρέπουν στι αστυνομικέ δυνάμει, να προστατεύουν την κοινωνία από το οργανωμένο έγκλημα, προστατεύουν και τα δικαιώματα στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε και την ε, ε, διατήρηση τη αναλογικότητα ω προ τον κίνδυνο. Αναφέρεται λοιπόν ότι μπορεί να γίνει αυτή η διατήρηση δεδομένων ε, για, κάποιου συγκεκριμένου, για την εντόπιση συγκεκριμένων κινδύνων τρομοκρατίας. Όμως δεν μπορούμε να διατηρούμε δεδομένα σε μεγάλο όγκο, όπως γινόταν στο παρελθόν. Και αυτή η απόφαση καταδεικνύει τα υψηλά πρότυπα ε, προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας που υπάρχει στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Και αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η απόφαση. Πλέον λοιπόν δεν ε, απαγορεύεται η μαζική ε, παρακολούθηση που παραβιάζει τα δικαιώματα τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση θα πρέπει να πληρεί πολύ συγκεκριμένα κριτήρια ε, τον, ε, τον, τα συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, το σκοπό της συλλογή των δεδομένων και πάντα πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση. Μετά την απόφαση τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια καλή ευκαιρία να τονίσουμε ε, προ το Συμβούλιο τη σημασία εξέβρεση συμφωνία για το κείμενο του πακέτου προστασία δεδομένων, ιδίω ε, στην οδηγία για την επιβόλη του νόμου. Θα πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε ε, υπό το φω και τη απόφαση. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη θέσει την τη γνώμη του και τώρα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η νομοθεσία. Ε, υπήρξε και έτοιμα ε, και ψήφισμα και από την ε, ΛΥΜΠΕ και τώρα θα πρέπει το Συμβούλιο να γνωρίσει την αξία του πακέτου αυτού, του νομοθετικού και να προχωρήσει ταχύτατα στην, στην διαπραγμάτευση για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Νιτφέλ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ την προσοχή στο εξής. Πολύ συχνά, έτσι και σήμερα, είναι από το Συμβούλιο. Απαράδεκτο. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο το ίδιο το 2005 πίεσε πάρα πολύ το Κοινοβούλιο για να υιοθετήσουμε βιαστικά αυτή την νομοθεσία σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και το να, τα αποτελέσματα. Ήταν κακή αυτή η νομοθεσία. Δεν θέλω να πω όπως αυτοί που καταψηφίζουν κάποια νομοθετήματα, σας το είπα εγώ, αλλά πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία. Δεν θα πρέπει τα δικαστήρια να ξεκάνουν αυτά που κάνουμε εμείς. Θα πρέπει εμείς να φτιάχνουμε ε, πολιτικές που να είναι νομικά βάσιμες. Αυτή είναι η ευθύνη μας ως πολιτικές. Όχι ε, πολιτικά τεχνάσματα, αλλά και νομοθετήματα νομικά βάσιμα. Νομίζω ότι αυτό που ζητάτε για μια, μια νέα οδηγία για την διατήρηση των δεδομένων είναι λιγάκι πρόωρο. Πριν περάσουμε και δώσουμε το μπαλάκι στην εθνική νομοθεσία, να σας πω ότι περιμένουμε μια πραγματική αξιολόγηση επί χρόνια. Και μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη δεν μας έδωσαν καθόλου στοιχεία, ούτε το παραμικρό στοιχείο, ότι χάρη σε αυτή την οδηγία, κύριε Βέμπερ, ο κόσμος είναι πιο ασφαλής. Ε, εξού και οι μαζικές παρακολουθήσεις. Και γι' αυτό και το δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτές οι μαζικές παρακολουθήσεις είναι δυσανάλογες. Πάμε τώρα στις επιπτώσεις. Καταρχά, θέλω να ακούσω την αξιολόγηση της Κομισιόν και θα ήθελα να μου πει ε, η Κομισιόν αν η αξιολόγησή τη είναι ομόφωνη για την επίπτωση στι εθνικέ νομοθεσίες. Από ό,τι ε, φαίνεται δεν ακυρώνται οι εθνικές νομοθεσίες αυτόματα. Και αυτό είναι περίεργο. Αυτό είναι περίεργο γιατί αν το δικαστήριο λέει ότι ας πούμε τα θεμέλια της οδηγίας είναι σαθρά ή δυσανάλογα, πώς η εθνική νομοθεσία που έχει ληφθεί για τη μεταφορά τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο να είναι σωστή. Όταν ξεκινήσετε, ε, θα ξεκινήσετε αντίστροφη διαδικασία επιπαραβάση αν τα κράτη-μέλη όπως η Ολλανδία δεν θέλουν να ακυρώσουν τις εθνικές νομοθεσίες, στην, ε, Ολλανδία δεν έχουμε καν συνταγματικό δικαστήριο. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την συνταγματικότητα των εθνικών νόμων τότε. Είναι δυνατόν οι εθνικοί νόμοι για τη διατήρηση των ε, δεδομένων να παραμείνουν ισχύ, άταν δεδομένα τα οποία συλλέγονται με βάση αυτού του νόμου χρησιμοποιείται α πούμε φερρυπίν από το Europol. Τι σημαίνει αν η Europol ε, συνεχεία με τη σειρά τη και αυτή παραβιάζει το δίκαιο. Εάν οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών απλώ αρνούνται να συνεχίζουν να συλλέγουν και να διατηρούν τα δεδομένα με βάση τι εθνικές νομοθεσίες. Τι γίνεται τότε. Επίση, τι πιστεύει ότι η Κομισιόν ότι είναι οι επιπτώσεις σε άλλα προγράμματα όπως το PNR, το SWIFT, το Eurodac ε, για τις πινακίδες αυτοκινήτων και οτιδήποτε άλλο. Η χρηματοδοτεί η Κομισιόν τη δημιουργία εθνικών συστημάτων για την ε, διατήρηση δεδομένων PNR σε 14 κράτη-μέλη. Μήπω είναι παράνομη αυτή η χρηματοδότηση, η Κομισιόν συμφωνείτε με αυτό. Και προ την Κομισιόν και στον κύριο Βέμπερ, τελευταίο ερώτημα. Ναι, σίγουρα θέλουμε να διατηρούμε ασφάλει του πολίτε μα, αλλά με αποτελεσματικού νόμου. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι αυτή η οδηγία ήταν αποτελεσματική. Η Κομισιόν τι σκέφτεται να κάνει, να έχει μια τελείω διαφορετική προσέγγιση, λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, πιο έξυπνα, ούτω ώστε να κρατήσουμε ασφαλεί πολίτε. Τι θα κάνετε. Δέχεστε από τον κύριο Βέμπερ, κυρία Ιντβέλτ, μία πλεκαρτα Κυρία Ιντβέλτ, ναι. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφε, εγώ παραμένω πιστός σε αυτό είπα. Είπα ότι υποστήριξα αυτό ότι χρειαζόμαστε μια πραγματική ισορροπία. Το ερώτημα το οποίο έχω σε εσά, αν δεν υπάρξει καμία νέα πρόταση από την Κομισιόν και δεν είπατε αν θέλετε μια πρόταση όχι, τότε ισχύουν τα εθνικά πρότυπα. Αν δείτε το βρετανικό μοντέλο, λιγότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θέλετε λοιπόν περισσότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ή όχι. Θέλετε μια νέα πρόταση Κομισιόν ή όχι. Κύριε Βέμπερ, το πρόβλημα είναι το αντίθετο ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είναι απαράδεκτο τα κράτη-μέλη να μην ακυρώνουν την, τους εθνικούς νόμους εφόσον παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό που προτείνετε εσείς είναι ξέπλυμα της πολιτικής. Ναι, εντάξει, να κρατήσουμε ασφαλή τους πολίτες μας, σωστό. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε. Έχουμε νόμους που βοηθούν προς αυτό, προς τη διατήρηση της ασφάλειας. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε αποδεικτικά στοιχεία και να με πείσετε, κύριε Βέμπε, εσείς που θέλετε τι μαζικέ παρακολουθήσει, ότι αυτή η οδηγία βοήθησε. Και αν ακούσατε προσεκτικά, εγώ είχα πει ε, προς την Κομισιόν, Κομισιόν, θα κάνετε προτάσεις εντελώς καινοφανείς, έξυπνους νόμους που θα προστατεύουν τους ανθρώπους και θα σέβονται παράλληλα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξηθεί το φαινόμενο του big data και δεν μπορούσε να γίνει λογικός διάλογος με ε, την ε, αστυνομία, την δικαιοσύνη και την πολιτική της δεξιάς. Διατηρούσαμε τα πάντα και η απόφαση του δικαστηρίου, ας μην υπάρχει παρανόηση, ε, λέει ουσιαστικά ότι δεν θα πρέπει ποτέ να έχει υπάρξει η νομοθεσία αυτή για την μαζική διατήρηση δεδομένων. Οτιδήποτε αφορά αυτή την πολιτική θα πρέπει να αναθεωρηθεί και μάλιστα γρήγορα το PNR κατά τη γνώμη μου μαζί με τις ΗΠΑ ε, πρέπει να έχει καταρρεύσει ουσιαστικά και το PNR με τον Καναδά, με την Αυστραλία και την Νότιο Κορέα ε, και οι, ε, οι ε, αποφάσει τη Επιτροπή για χώρε όπω η δική μου για την διατήρηση εθνικού προγράμματο διατήρηση στοιχείων των επιβατών και για το SWIFT. Θα πρέπει να σταματήσει επιτέλου η μεταβίβαση των δικών μα τραπεζικών στοιχείων στι ΗΠΑ, γιατί αυτό είναι κάτι το παράνομο. Οι Βρετανοί κατάσκοποι παρακολουθούν τις δικές μας συνομιλίες, τις αντιγράφουν τα δεδομένα μας και τα διατηρούν. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Επιτέλους, υπεράσπιση των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε διαφορετική προσέγγιση και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ε, μεθόδους ε, ε, ανείχνευση και εντοπισμού, όπω είναι το quick freeze. Ε, δεν υπάρχει τώρα νομοθεσία, πρέπει να υπάρξει όμω. Και σίγουρα, αν εμεί περιμένουμε τι κυβερνήσει μα, θα περιμένουμε. Ε, για, για παράδειγμα, στη χώρα μου χρειαζόμαστε ακόμα 8 εβδομάδε. Εγώ καλώ ε, τι ε, αντίστοιχε εταιρείε να σταματήσουν τώρα την καταγραφή των προσωπικών μα δεδομένων και οι κυβερνήσει μα το έχουν χάσει. Επομένω, α είμαστε λοιπόν ε, ανυπάκουοι σε αυτή την περίπτωση, γιατί αλλιώ θα το κάνουν οι πολίτε μα. Κατά του φόβου λοιπόν μιλώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε με την κυρία Έρνστ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη διατήρηση στοιχείων έχει μια πολύ μεγάλη σημασία διότι ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μια απόδειξη σε αυτή την απόφαση ότι λειτουργεί η προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είναι φανερό ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται για αυτά τα δικαιώματα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν αυτούς τους ακτιβιστές από την ε, Αυστρία, από την Ιλλανδία και όλους αυτούς που υποστήριξαν αυτή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της κράτησης δεδομένου. Η απόφαση αυτή είναι σαφής και τονίζει ότι η οδηγία αυτή είναι μια λαθασμένη οδηγία και πρέπει να αρθεί και αναδρομικά η ισχύ τη. Δεν είναι λοιπόν έγκυρη. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Λέει το δικαστήριο ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία χρησιμοποίηση του κοινού συμφέροντος για να υποστηριχθεί η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως, όπως σε αυτή την οδηγία. Δεν υπάρχει καμία λοιπόν άμεση σύνδεση κύριε Βέμπερ μεταξύ της κράτησης δεδομένων και κάποιας οποιασδήποτε απειλής όπως από την τρομοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες απαραίτητοι περιορισμοί, όπως λέει η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων. Και εμεί ζητούμε όλες οι οδηγίες, όλοι οι κανονισμοί που περιλαμβάνουν τέτοιες ρήτρε για συλλογή δεδομένων να εξεταστούν και πάλι. Ο της συλλογής δεδομένων, η Europol, η Eurodac, όλες αυτές οι συμφωνίες που συλλέγουν στοιχεία ακόμα και από πρόσφυγες. Αυτό είναι μια έκφραση ρατσισμού. Θυμίστε, το SWIFT, το PNR, τις συμφωνίες αυτές με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σήμερα την ευκαιρία για να κάνουμε σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό PNR. Και αυτό το τονίζει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να άρουν οποιαδήποτε ε, διάταξη που έχει να κάνει με τη συλλογή τη δεδομένων, γιατί αυτή είναι αντίθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ζητούμε από την Κομισιόν επίσης να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξουν διαδικασίες επί παραβάση κατά των κρατών που δεν κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να ακυρώσουν αυτήν την ε, κράτηση δεδομένων. Λοιπόν, είναι πια κάτι το οποίο το έχουμε καταδικάσει, τη μαζική αυτή παρακολούθηση των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει σαφή θέση για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βος έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Αξιότιμη κυρία Επίτροπος. Είναι πολύ θετική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί διευκρινίζει ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η κράτηση δεδομένων και σε ποιες όχι. Έτσι διασαφηνίζει την οριοθετική γραμμή. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι το μόνο ε, συμπέρασμα που παίρνει κανείς από την απόφαση του Συμβουλίου είναι ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να έχει καμία πρόταση για κράτηση δεδομένων και βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί κίνδυνοι και ούτε μπορούμε να δεχτούμε να συνεχιστούν ε, καταστάσεις οι οποίες έχουν σωστά αναφερθεί σε σχέση με το SWIFT για τα κενά ασφαλείας. Αυτός δεν είναι ένας λόγος όμως να μην υπάρχουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ και ένα καθεστώς σε σχέση με την κράτηση δεδομένων. Πέραν του δικαιώματος στην ελευθερία υπάρχει και το δικαίωμα στην ασφάλεια. Αναφέρεται στο άρθρο 6 της ε, Χάρτας Ανθρωπινών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί η σοβαρή εγκληματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ούτε το άλλο συμπέρασμα που προτείνω ορισμένοι ότι επειδή η ποινική δίωξη είναι αποκλειστικό δικαίωμα του έθνους κράτους να μην γίνονται ενέργειες οι οποίες αλλιώς δεν θα μπορούσαν να διωχθούν καθόλου. Όταν λοιπόν δεν φτάνει ένα κράτος για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα, λένε ορισμένοι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία δίωξη. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα αντίθετο με την έννοια του δικαίου, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα των διοκτικών αρχών να προχωρήσουν σε δίωξη ακόμα και να χρησιμοποιήσουν όλα τα τεχνικά εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεσή τους. Εμείς ως νομοθέτες λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας, δηλαδή ένα επίπεδο ασφάλειας το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και επομένω, εδώ είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνη των πολιτών μα στι διοκτικέ αρχές, στις δικαστικές αρχές, στην αστυνομία αλλά εν γέννη σε όλο το κράτος δικαίου. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι και τα θεμητά συμφέροντα των θυμάτων εγκλημάτων τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την ισορροπία που ανέφερε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών για την προστασία των δεδομένων τους, αλλά και τα δικαιώματά τους να διαλευκαίνονται τα εγκλήματα και να υπάρχει η δικαιοσύνη για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών και δεν πρέπει να τους λέμε ότι δεν διαλευκάθηκε μια περίπτωση γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία. Κύριε Βόση, υπάρχει μια μπλε κάρτα, υπάρχουν περισσότερες από μια μπλε κάρτε, μάλλον επειδή έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Σας παρακαλώ να θέτετε μόνο ερωτήματα, κυρία Ιντφέλτ. Ε, Η κυρία Έρστ, μάλλον, συγγνώμη. Αγαπητέ συνάδελφε. Η κυρία Ιντφέλτ, υπονοείται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορείτε παρακαλώ... Όχι, Πράγματι, θέλω να μου απαντήσετε. Μπορείτε επίσης, σας παρακαλώ θερμά, μετά από 8 χρόνια που σας το ζητάμε, μπορείτε να μας δώσετε αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της μαζικής ε, ε, αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι μόνο ε, δεδομένα τηλεπικοινωνιών που έχουν αποθηκευθεί, κάθε είδους δεδομένα που δεν έχουν αποτρέψει μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Κόβω το μικρόφωνο της ομιλήτριας άλλο ερώτημα από την κυρία Ένστ. Και εμένα το ερώτημά μου κινείται προ την ίδια κατεύθυνση. Αν κοιτάξετε αυτή την ε, απόφαση το σημείο 95, 59 συγγνώμη, είναι σαφές ότι η συλλογή δεδομένων ε, δεν μπορεί κανείς με αυτά τα στοιχεία να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία. Αυτό το βλέπετε λοιπόν μέσα στο σκεπτικό της απόφασης και εσείς πώς λέτε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς συλλογή δεδομένων οι διοκτικές αρχές και δεν συλλέγουν τέτοια δεδομένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όλα, όλες αυτές οι συνδέσεις δεδομένων δεν μπορούν να ισχύουν και να υπάρχουν όταν δεν έχουμε συλλογή δεδομένων και τα δικαστήρια δεν μπορούν να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει η χώρα ένα αδίκημα, ένα έγκλημα. Προφανώς μπορεί να προχωρήσει κανείς σε αντιμετώπιση ε, εγκλημάτων, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να ξέρει κανείς ενδελεχώς τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν πρόκειται λοιπόν για, την, για τον εμποδισμό μονάχα αδικημάτων, αλλά για την δυνατότητα δίωξης με πλήρη χρήση αυτών των σημείων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον νόμο και τα θεμελιώδη δικαιώματα και όχι όπως ορισμένοι ε, νομοθέτες μπορεί να το αντιμετωπίζουν τι πρέπει να κάνει περισσότερο το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει λοιπόν να σεβαστεί την ελευθερία των μεν και των δε αλλά χωρίς να ξεπεράσει τα όρια τα οποία θέτει το δίκαιο. Ο κύριος Λόπες Αγγελάρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μία εβδομάδα και κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου αποφάσισε ότι είναι ασύμβατη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οδηγία του 2006 για την τήρηση δεδομένων. Το είπε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος ήταν σαφές, σαφής. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι αυτό είναι ένα θαυμάσιο νέο για 500 εκατομμύρια πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για νομικού λόγου, αλλά κυρίω για πολιτικού και δημοκρατικού λόγου. Για λόγου νομικού, γιατί είναι πάρα πολύ σαφή και υποδειγματική αυτή η απόφαση και τονίζει τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ελευθερίες των πολιτών. Και λέει ότι η οδηγία αυτή δεν είχε την αναλογικότητα η οποία να δικαιολογεί την συλλογή και κράτηση αυτών των δεδομένων. Απλώς χρησιμοποιούσε αυτήν την έννοια ότι συλλέγουμε όλα τα δεδομένα μήπως μας χρειαστούν κάποια στιγμή. Αλλά αυτό είναι αντίθετο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για σε ό,τι αφορά. Λοιπόν, αυτή την απόφαση χρησιμοποίησε σαν βασικό στοιχείο, ως στοιχείο παραγόγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επομένως, έπαιξε ένα ρόλο συνταγματικού δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστήριο, ελέγχοντας τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτή τη οδηγία. Αυτό δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό από νομική άποψη αλλά και από κοινωνική, από πολιτική και από δημοκρατική άποψη. Γιατί αυτοί οι οποίοι θέλουν να αναγάγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ατέρμονη συζήτηση για την διακυβέρνηση του ευρώ, την χρηματοπιστωτική κρίση, την διαχείριση της εσωτερικής αγοράς θέλουν να την κάνουν μονάχα μια οικονομική και νομισματική ένωση. Όλοι αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει και με τις ελευθερίες των πολιτών και τα δικαιώματα των πολιτών και πρέπει να καταλάβουν ότι η απόφαση αυτή ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών. Και ενώπιον των εκλογών της 25ης Μαρτίου θα πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε περισσότερο και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων στην ιδιωτική μορφή και την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Σε αυτό είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθέτη και ως υποστηριχτή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνεχίζει ο κύριο Αγγελάρ χωρί μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Λόπε Αγγελάρ. Σα παρακαλώ να παραμένετε μέσα στο χρονογράφηση γιατί έχουμε καθυστερήσει. Κύριε Λάντφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια απόφαση ορόσημα για την προστασία δεδομένων για τη ιδιωτική σφαίρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν αυτή και θέτει όρια για το τι μπορεί να γίνει δεκτό ε, σε ό,τι αφορά του περιορισμού ε, των ελευθεριών προ την αναζήτηση ασφάλεια. Θα το συζητούμε εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον τα 15 χρόνια που εγώ είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το σύστημα αυτό έχει γίνει όλο ένα και πιο περίπλοκο ε, σε μια εποχή ε, και διαδικτυακής ε, διατήρησης δεδομένων και επικοινωνίας. Εγώ είμαι αντίθετη με την οδηγία του 2005 και αντιτάχθηκα σε αυτή την οδηγία βάσει και των όσων είπε και ο εισηγητής Αλεξάλγορα όπως αναφέρθηκε, είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολιτικής, ε, ξεπλήματος πολιτικής, όπως είπε και η κυρία Ιντφέλτ. Και το Μήνο Βασίλειο ήταν στο Συμβούλιο, στην Προεδρία του Συμβουλίου, που μετά έγινε ήταν ε, και υπουργό ε, των εργατικών, Charles Clark. Δεν κατάφεραν λοιπόν να περάσουν μία υποχρεωτική ε, διατήρηση δεδομένων στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Δεν υπήρχε δηλαδή Βρετανικός νόμος για αυτό το ζήτημα. Τι γίνεται λοιπόν, περνάει μέσα από τις Βρυξέλλες και με την συνενοχή των Σοσιαλιστών και του ΕΛΚ. Ήταν ένα ε, απαράδεκτο παράδειγμα ξεπλήματος πολιτικής. Ε, και ε, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δείχνει ότι αυτή η διατήρηση δεδομένων είναι μια αδικαιολόγητη και υπέρμετρη ε, παραβίαση δικαιωμάτων, ε, το οποίο εμεί το είχαμε εντοπίσει το 2005. Πράγματι, θα πρέπει τα κρατημέλη να αναθεωρήσουν τι εθνικέ του νομοθεσίε για να ε, συμμορφούνται με την απόφαση και Ιδάλω, ε, σίγουρα θα το πράξουν τα εθνικά δικαστήρια. Οι κυβερνήσει σίγουρα θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύουν του πολίτε του από το σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Όμω, ε, η άμεση προσφυγή στην ε, μαζική κατασκοπία και παρακολούθηση χωρί βάσιμε υποψίε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η μαζική κατασκοπία λοιπόν και παρακολούθηση των πολιτών μας μαζί με την ε, αδικαιολόγητη παρακολούθηση με ελλειπή εποπτεία ε, και λογοδοσία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε. Δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι και επικαλούμαστε την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να αιτιολογήσουμε τις ε, δυσανάλογες επιπτώσεις και περιορισμό της ελευθερίας υπήρξε συγκεκριμένη επίκριση για την έλλειψη προϋπόθεσης δικαστική απόφαση πριν περάσουμε σε διατήρηση δεδομένων. Το δικαστήριο λοιπόν ε, υποστηρίζει και περασπίζεται τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Και ε, απαγορεύει πλέον αυτή τη μαζική διατήρηση δεδομένων. Και ελπίζουμε έτσι να τεθεί ένα τέλος αυτή τη δεκαετία μαζικής παρακολούθησης. Εγώ προσβλέπω με ανυπομονησία να δω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για το PNR και για τη συμφωνία SWIFT. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα που οδηγήσαμε στην διερεύνηση των πρακτικών και από τον κύριο Μωράες ο οποίος εξηλαιώθηκε ε, για την ψήφο του 2005. Εμεί ζητούμε απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα. Διέκοπτε το, ερώτημα, το μικρόφωνο τη ομιλήτρια. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε με την κυρία Λατσέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Η απόφαση τη 8 η Απριλίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πραγματικά κάτι το οποίο ουσιαστικά απελευθερώνει από ένα μεγάλο βάρο τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε και η συνάδελφό μου, η κυρία Σαργεντίνη, έδρασε εναντίον του φόβου και αυτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον φόβο και υποστήριξε την ελευθερία και τι ελευθερίε των πολιτών. Γιατί υπήρξε αυτή η οδηγία και πώς καταρρίφθηκε. Πρέπει να σας την πετιμήσω. Ο Άλμπερ Στάινχάουρ από το δικό μου κόμμα αποφάσισε να προσφύγει στο Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο με μια προσφυγή κατά της νομοθεσίας για την κράτηση δεδομένων. Αυτό κράτησε λίγους μήνες και σύντομα είχε μαζί του σχεδόν 12.000 υπογραφές που υποστήριξαν την ενέργεια αυτή. Ήταν η μεγαλύτερη συνταγματική δίκη που έγινε στη δημοκρατία της Αυστρίας ενέκρινε λοιπόν ως παραδεκτή την προσφυγή αυτή το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο γιατί θεώρησε ότι υπάρχει πρόβλημα παρέμβαση στην ε, ιδιωτική σφαίρα χωρίς να υπάρχει αναλογική, αναλογικότητα με τους στόχους, δηλαδή την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Δεν υπήρξε λοιπόν αναλογικότητα των μέλων, των ε, μέσων που χρησιμοποιούνται θεώρησε ότι υπάρχει μια σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας η οποία δεν είναι παραδεκτή. Χαίρομαι λοιπόν που το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο έθεσε προδικαστικό ερώτημα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υποστήριξε ότι πράγματι υπάρχει αυτό το θέμα της αναποτελεσματικότητας και όχι μόνο της ε, έλλειψης αναλογίας. Με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει ότι τα, η εθνική νομοθεσία για τα θέματα αυτά πάβει να ισχύει πλέον και δεν είναι έγκυρη. Κυρία Βεζιά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία που ακύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 8 Απριλίου υιοθετήθηκε μετά την, τις τρομοκρατικές επιθώσεις στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο. Ε, Φυσικά, λόγω της δημοκρατία πρέπει να πάρουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό, αλλά όχι όπως να είναι. Το δικαστήριο υπενθύμησε σωστά ότι ο νομοθέτης πρέπει να σεβαστεί τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές αρχές που είναι η αρχή της αναλογικότητας. Αυτή η οδηγία είχε υποχρεώσει δυσανάλογα του παρόχου υπηρεσιών και τους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ να διατηρούν γενικά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την προέλευση, την, την, τον προορισμό, την ώρα, το είδος της επικοινωνίας, την ε, τεχνολογία που χρησιμοποιείται, την ε, θέση επίσης. Είναι μια γενική δηλαδή ε, παρακολούθηση μαζικού χαρακτήρα και ξέρουμε μετά την Ερευνητική Επιτροπή για άλλες υποθέσεις ότι αυτή δεν είναι η καλή μέθοδος μόνο οι στοχευμένες προσεγγίσεις είναι σωστές για το δικαστήριο. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να βρούμε τη σωστή και διαβόητη ισορροπία. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει στην εποχή εκείνη είχαν καταγγείλει αυτή την οδηγία, ακόμα και τη στιγμή που μεταφερόταν στην εθνική νομοθεσία. Πολλά κράτη-μέλη, μάλιστα, άργησαν να την ενσωματώσουν στην εθνική του νομοθεσία και πολλά σταγματικά δικαστήρια σε πολλά κράτη-μέλη είχαν κρίνει ότι η οδηγία είναι ασύμβατη με το Σύνταγμα διαφόρων κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πίστευε ότι η οδηγία αυτή ε, υπησερχόταν με τρόπο απαράδεκτο ε, στην ιδιωτική σφαίρα και στα προσωπικά δεδομένα ε, σε ό,τι αφορά λόγω του εύρους συλλογής των δεδομένων, τη διατήρησή τους κτλ. Το δικαστήριο απλώς ε, επαναλαμβάνει τα παράπονα που πάρα πολλοί από εμά επαναλαμβάναμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και τα κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει αυτήν την οδηγία θα πρέπει να αναστείλουν την εφαρμογή της. Εάν γίνει αναθεώρηση θα πρέπει να είναι στο ύψος ε, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Κομισιόν ξέρει ότι σε κάποιους τομείς, κυρίως οικονομικούς, το να τη σεβαστεί στην την νομολογία του δικαστηρίου είναι σωστό και πρέπει να σέβεται επίσης και την νομολογία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ελπίζω να σταματήσει αυτή η ιστορία με την καταστολή που μας έχει ζώσει τα τελευταία χρόνια. Όταν υιοθετήθηκαν οι συμφωνίε SWIFT, PNR, η SEFAR με τι ΗΠΑ, υπήρξε πρόβλημα. Όλε οι διεθνεί συμφωνίε σε αυτό το τομέα θα πρέπει να ανασταλούν, καθώ και η σχετική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, θα ευθυγραμμίσουν τα έργα και τα λόγια του και οι Ευρωπαίοι πολίτε θα χαρούν γιατί πρέπει οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν σεβαστέ. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κέλλη είναι ο επόμενο ομιλητή. Όσοι ήταν υπέρ αυτής της οδηγίας, δεν είναι εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαστήριο κοίταξαν το πράγμα ανεξάρτητα και πήραν μία απόφαση την οποία θα πρέπει εμείς να δεχτούμε ως χαρμόσυνο νέο. Ε, ξέρετε για την απόφαση αυτή που αφορούσε την εταιρεία Digital Rights Ireland, καθώς και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας. Δεν χρειάζεται κανένας να ανησυχήσει, γιατί το πρώτο σημείο που αφορά το τι θέλουμε να πετύχουμε είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι νόημα έχει να τα απαιτούμε σε όλο τον πλανήτη αν εμείς δεν τα έχουμε. Με αυτή την απόφαση ξεκαθαρίζεται ότι η καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και τελικά η δημόσια ασφάλεια λέει το δικαστήριο με την υιοθέτηση της οδηγίας αυτής η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης υπερεύει α, τις υποχρεώσεις του και την αρχή της α, αναλογικότητας. Ε, παρεμβαίνει σοβαρά αυτή η οδηγία στα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν οριθετείται αρκετά αυτή η οδηγία ούτω ώστε αυτή η παρεμβολή στα θεμελιώδη δικαιώματα να περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να την κοιτάξουμε, να εξασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε την αντικαταστήσει δεν θα ξεπερνάει τα όρια και μην ξεχνάτε ότι σήμερα όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το ίντερνετ και θα πρέπει να ξέρουν ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή. Και όσοι ε, εξασφαλίζουν ε, την εφαρμογή του νόμου, οι διοκτικές αρχές κτλ. θα πρέπει να σέβονται την νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Γκίγιόμ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο όμω πάντα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή τη ε, συζήτηση και του διαλόγου και την προστασία δεδομένων. Ε, με την απόφαση τη περασμένη εβδομάδα ε, φαίνεται ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη μάχη. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την νομιμότητα των ε, στόχων ε, της οδηγίας, τη ε, διατήρηση των προσωπικών δεδομένων, όμως εκτίμησε ότι η συστηματική διατήρηση και χωρίς εξαιρεσει αυτών των δεδομένων από όλου του Ευρωπαίου παρόχου για αόριστη διάρκεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επομένω, πρόκειται για σημαντική παραβίαση τη ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων. Οι αδυναμίε του κειμένου που υιοθετήθηκε το 2005 σε ένα ιδιαίτερο ε, πλαίσιο μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει μα είναι γνωστό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μήπω έχει φτάσει στα ε, όρια τη ε, σε αυτή την εκτίμηση. Επίση, θεωρούμε ότι πρόκειται για κάτι παροχημένο ε, μέσα στην προσέγγιση του Big Data ε, και τη νέα πραγματικότητα που επιτρέπει την ε, συλλογή δεδομένων χωρίς κανένα περιορισμό. Επομένω, ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να συναγάγουμε ότι ε, δεν είχαμε μόνο ε, εύρω στους κανόνες για την προστασία δεδομένων, θα έπρεπε να υπάρχει, είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ για να διασφαλίσουμε την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και την στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Φαίνεται ότι υπήρξαν πολύ σημαντικές καταχρήσεις των δημοκρατικών ελευθεριών Εάν το σοβαρό έγκλημα και η τρομοκρατία είναι κάτι το οποίο μα απασχολούν ακόμα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αυτό σε βάρο των δημοκρατικών αληθινών των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν μπορεί να γίνει μόνο σλόγγαν. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό περιμένουμε από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να προτείνει ε, νέο κείμενο. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Βίξτρομ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων και είναι απολύτω ε, σαφή αυτή η απόφαση. Η νομοθεσία που υιοθετήθηκε στα κράτη-μέλη μα θα πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί. Και έτσι η διατήρηση δεδομένων θα πρέπει να συμβαίνει μόνο εντός ε, συγκεκριμένων και εξαιρετικά σαφών περιορισμών βάσει αυτή τη απόφαση. Και η αποθήκευση των δεδομένων όπως συμβαίνει τώρα, δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις μας ελευθερίες και τα δημοκρατικά μας δικαιώματα βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ επικροτώ τη σαφήνεια της απόφασης του δικαστηρίου Έχουμε θέσει πολύ ψηλά τον τύχη, πύχη συγγνώμη, με τα κράτη-μέλη όταν μιλάμε για δημοκρατικέ ελευθερίε και βεβαίω και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει το ίδιο και τα δικαστήριά τη. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια ευκαιρία να βελτιώσουμε την νομοθεσία μα. Η συλλογή ηλεκτρονικών δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Δεν θα πρέπει να γίνεται όταν δεν υπάρχουν υποψίε. Επίση, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία, την εφαρμοστική νομοθεσία στα κρατη θα πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου κατά την αναθεώρηση του ιστορικού του εθνικού δικαίου. Και τέλο, ένα ακόμα ερώτημα που ανακύπτει εάν θα γίνεται, αν θα θεσμοθετήσουμε νομοθεσία μέσω οδηγιών ή κανονισμών. Οι κανονισμοί εφαρμόζονται άμεσα ε, στα κράτη-μέλη, ενώ οι οδηγίε ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία. Η διαδικασία είναι δύσκολη και πρέπει να ε, ε, ελέγχουμε αν γίνεται η διαδικασία ως, όπως πρέπει. Καλύτερα θα, θα καλό θα ήταν να εργαζόμαστε με κανονισμού ε, στο μέλλον και όχι με οδηγίε. Και, ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω το γεγονό ότι η Επιτροπή θα αποζημιώσει τη Σουηδία, η οποία κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο στο παρελθόν, γιατί θεωρήθηκε ότι η Σουηδία δεν εφαρμόζει ε, όπως θα έπρεπε την οδηγία. Επομένω, καλό είναι που αποζημιωνόμαστε. Ευχαριστώ. Κύριε Σουλέτερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονό ότι 8 χρόνια μετά από την ψηφοφορία που έχει γίνει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο, χάρη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορέσαμε να έχουμε ένα πραγματικό μια πραγματική αντιμετώπιση. Γιατί αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ηλίθια και ουσιαστικά σπατάλησε πάρα πολλά λεφτά. Αν είχαμε ακούσει αυτά που είχε πει ο αρμόδιος για τα προσωπικά δεδομένα, δεν θα είχαμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δυστυχώ τον αγνοήσαμε τώρα. Ευτυχώ δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το δικαστήριο. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ότι όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την απόφαση του δικαστηρίου. Οποιαδήποτε νομοθεσία η οποία είναι αντίθετη με αυτήν την απόφαση θα πρέπει να ακυρωθεί. Ένα άλλο σημείο που θέλω να δείξω είναι και το εξή. Η αποτελεσματικότητα αυτής μεθόδου ήταν μηδενική. 0,006% όπως έδειξε μια γερμανική μελέτη βοηθήθηκαν από την κράτηση αυτών των δεδομένων. Τίποτα, αυτό δεν μετράει. Δεν μπορέσαμε να εμποδίσουμε με αυτά τα μέτρα κανένα έγκλημα και συγχρόνως ήταν μια τόσο μεγάλη παραβίαση ιδιωτική μα ζωή. Κοιτάξτε όμω τι λέει η απόφαση, γιατί το δικαστήριο επικρίνει ορισμένε αρχέ. Την χίδινη συλλογή δεδομένων που που καλύπτουν ευαίσθητες πληροφορίες για κάθε πολίτη. Εκεί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της παράνομης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα που είναι ένας μεγάλος δυνητικός κίνδυνος. Αυτό εφαρμόστηκε στην περίπτωση του PNR, του SWIFT και εφαρμόζεται και σε εθνικές νομοθεσίες όπως η νομοθεσία FRA της Σουηδίας. Γι' αυτό θέλουμε να παροτρύνουμε την Κομισιόν να αναθεωρήσει και να <clears throat> εξετάσει όλες τις μορφές νομοθεσίες που βασίζονται στην κράτηση δεδομένων και που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι παράνομες επί τη βάση απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για να υπάρξει αυτή η ακύρωση κάθε νομοθεσίας που είναι αντίθετη με την απόφαση. Ο κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση δεν μπορούσε να έρθει σε καλύτερη χρονική στιγμή μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχει παγκόσμια συνειδητοποίηση ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μαζική ε, αντιμετώπιση παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων έχουν αποκαλυφθεί από τον Edward Snowden η μαζικότητα όλων αυτών των ε, ε, συλλογών δεδομένων. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πολύ σωστό αυτό που έκανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είναι ηρωνικό αυτό που λένε πολλά μέλη του Κοινοβουλίου εδώ, γιατί πριν από λίγα χρόνια αυτοί είχαν επιτρέψει να περάσει αυτή η οδηγία και λένε τώρα ναι, τι καλά που τα έκανε το δικαστήριο και εξακολουθούν να λένε ότι πρέπει να αγωνιστούμε αντίον της τρομοκρατίας, είναι σαν να λένε ότι δεν δέχονται αυτή την απόφαση. Έχουμε <clears throat> ουσιαστικά με την απόφαση αυτή είχαμε ιδιωτικοποιήσει τον μεγάλο αδελφό. Οι, ε, οι πάροχοι του ίντερνετ, οι τηλεφωνικές εταιρείες ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι μας κατασκοπεύαν και κρατούσαν τα δεδομένα μας για δύο χρόνια. Ποιο θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μονάχα οι ακτιβιστές στην Ιρλανδία και την Αυστρία που αντιμετώπισαν αυτό το θέμα, που αγωνίστηκαν, που το φέρανε στην Ιρλανδία στα δικαστήρια χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα να διαμφισβητήσουν την νομιμότητα αυτής της νομοθεσίας στην Ιρλανδία. Και τώρα δεν έχει τελειώσει εξάλλου γιατί είναι όλες αυτές οι χώρες οι οποίες έχουν περάσει εθνική νομοθεσία πρέπει να υπάρξει διαφυσβήτηση στα δικαστήρια από τη βάση, από τους απλούς πολίτες. Δεν χρειάζεται γιατί η Κομισιό θα μπορούσε ήδη να πει ότι αυτή η νομοθεσία είναι απόλυτη παράνομη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η νίκη δεν θα <clears throat> ανατραπεί γιατί μερικά από τα σχόλια των μελών του ΕΛΚ και της εκπροσώπου της Κομισιόν στο παρελθόν είναι ανισχυτικά. Γιατί η, Κομισιόν, η εκπρόσωπος, Κομισιόν είπε ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στον αγώνα κατά του εγκλήματος και τη νομοκρατία. Και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό με την απόφαση του δικαστηρίου. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αντιδημοκρατικέ οδηγίε τύπου μεγάλου αδερφού από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως θα σταματήσετε πια να χρησιμοποιείτε τη δημοκρατία ω πρόσχημα για να παραβιάσετε την ιδιωτικότητα των πολιτών μα. Ο κύριο Βάιντεν Χόλτσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την συλλογή και κράτηση δεδομένων είναι μια πολύ σημαντική νομική πράξη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν <clears throat> υπάρχει μια ε, σημαντική χρησιμοποίηση της Χάρτας Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Είναι μια πραγματική ιστορική στιγμή. Έχει γίνει σαφές ότι η μαζική συλλογή δεδομένων και η κράτησή τους και η δημιουργία τεραστίων βάσεων δεδομένων δεν έχει οδηγήσει σε καμία ασφάλεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Ε, η εντύπωση ότι όλοι είμαστε με την εντύπωση ότι μας παρακολουθούν δεν αυξάνει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Και η νομολογία του δικαστήριου λοιπόν τονίζει ότι δεν μπορεί αυτή η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής να συνάδει με την χάρτα θεμελιωδεών δικαιωμάτων. Η έλλειψη λοιπόν μιας αναλογίας έγινε κάτι έγινε σαφής από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτά όμως καταδεικνύει ότι λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι και αυτή η απόφαση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια τροποποίηση των ε, αντιμετωπίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι οδηγίες οι οποίες θα ακολουθήσουν θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν ένα στοχευμένο χαρακτήρα δεν έχει νόημα η συλλογή των δεδομένων μέσα στι οδηγίε αυτέ. Και αν έχει κάποιο νόημα ούτω ή άλλω, αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Ευρωπαίο πολίτη. Πρέπει όμω η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον να σέβεται την ιδιωτικότητα των πολιτών, είτε είναι ε, για του τραπεζικού λογαριασμού στο SWIFT, είτε για τα δεδομένα του όταν ταξιδεύουν. Πρέπει πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλήσει τα απαραίτητα συμφέροντα. Δεν μπορεί λοιπόν από εδώ και πέρα να αναφέρεται κανείς σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί λοιπόν με χίδιν τρόπο να συλλέγονται και να κρατώνται προσωπικά δεδομένα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Χίρς. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το στικάκι να κρατώνται εκατομμύρια στοιχεία για συνδιαλέξεις Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή λοιπόν η αλόγιστη συλλογή και κράτηση δεδομένων έχει φτάσει επιτέλους σε ένα τέλος. Αυτό αφορά όλους μας. Μας θέτει αυτή η διαδικασία όλους κάτω από μια συλλήβδην υποψία. Δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει πρέπει η Κομισιόν να ζητήσει συγγνώμη από τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί επί χρόνια μας έχει σπιουνάρει και έχει κρατήσει τα προσωπικά μας δεδομένα χωρίς αυτό να οδηγήσει σε τίποτα σε επίπεδο προστασίας. Είναι κάτι το οποίο μας σοκα... σοκάρει και το αυτό το οποίο μας εντυπωσιάζει είναι ότι οι συντηρητικοί συνάδελφοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θέλουμε μια νέα οδηγία της Κομισιόν για την κράτηση δεδομένων. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου. Είναι έτοιμοι να καταπατήσουν πάλι τα δικαιώματα των πολιτών συγχέοντας όλα αυτά με την καταπολέμηση του, ε, <clears throat> της τρομοκρατίας και της ε, εγκληματικότητας. Η η αρμόδια υπουργό στη Γερμανία έχει ε, εμποδίσει την προστασία των πολιτών. Τώρα λέει ότι η αστυνομία δεν χρειάζεται αυτή την ε, συλλογή δεδομένων. Και δεν χρειαζόμαστε πράγματι ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Κυρία Ζήπελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει ακυρώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την συλλογή δεδομένων. Πρέπει να υπάρξει προστασία των πολιτών, αλλά η ελευθερία και τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίας πρέπει να ισχύουν παντού. Δεν αντιμετώπισε το δικαστήριο μόνο το χρόνο και άλλες λεπτομέρειες. Τόνισε ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να συλλέγει και να κρατά δεδομένα όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν συνάδει με βασικές νομικές αρχές όπως το τεκμήριο αθωότητος των πολιτών. Μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παραμένει μονάχα ένα ερώτημα. Θα κάνει μια νέα πρόταση κομισιόν ή αυτή η διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων δεν υπάρχει πια. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα όμως. Αν αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν ισχύει ακριβώ και το ίδιο για τη μεταγραφή του στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. <clears throat> Μήπω θα πρέπει να αντλήσουμε λοιπόν το συμπέρασμα ότι όλε οι εθνικέ μεταγραφέ στο εθνικό δίκαιο δεν έχουν πια νομική αξία. Και αυτό ισχύει βέβαια και για όλα τα δεδομένα όπω είναι από το SWIFT, το Passenger Name Record κτλ. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν τη συζήτηση που έχει γίνει για την ε, ε, χρήση δεδομένων από τις μυστικές υπηρεσίες των δεδομένων των ε, επιχειρήσεων είναι φανερό ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πού πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε πώς θα προστατεύσουμε τις προσωπικές ελευθερίες και τα δεδομένα και στον ψηφιακό κυβερνόχωρο. Χρειαζόμαστε να έχουμε μια νομοθεσία η οποία θα σέβεται τις δημοκρατικές αρχές και τις αρχές του κράτους δικαίου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περιμένουμε την κυρία Γκόμες. Ήρθε. Την περιμένουμε ή όχι. Όχι. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριο Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, στην απόφασή του το δικαστήριο είπε ότι η οδηγία αποτελεί απίστευτη παρεμβολή στα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, ε, δεν σέβεται την ιδιωτική σφαίρα και τα προσωπικά ε, προσωπικό χώρο. Συμφωνώ. Το να κρατούμε αδικαιολόγητα και για όσο χρονικό διάστημα αυτά τα δεδομένα παράδεκτο. Μία αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής επιβάλλεται και επομένως πολλών άλλων νομοθετημάτων που εμπνεύστηκαν την οδηγία. Ε, το PNR, το SWIFT, όλα αυτά που ακούστηκαν, που συλλέγουν ε, καταχρηστικά δεδομένα εις βάρος των πολιτών, των ε, ατομικών ελευθεριών, του σεβασμού της ιδιωτικής σφαίρας. θα πρέπει να αμφισβητήσουμε ένα τμήμα αυτών των συμφωνιών. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείες το δικαστήριο υπενθύμησε αυτούς που δεν μας πίστευαν ότι η προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδου σημασίας αξία στην, ε, ε, στις κοινωνίες μας και σε ό,τι αφορά την ε, ελευθερία 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ο επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέει ο Σέγγστρομ, είπε ότι είναι παράνομη αυτή η οδηγία, είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι άκυρη και πρέπει να αποσυρθεί. Ε, υπάρχουν όμως και πολλές εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζουν στο εθνικό δίκαιο αυτή την οδηγία και δυστυχώς αυτές ακόμα ισχύουν. Κυρία Επίτροπε, έχετε ευθύνη απέναντι στα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, κύριε Επίτροπε, τι θα κάνετε εσεί, ούτω ώστε να εξασφαλίσετε ότι αυτέ οι χώρε ανακαλούν αυτή την νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. Ε, στη δική μα χώρα, Φερρυπίν, τη Σουηδία. Ένα ε, καλό παράδειγμα είναι. Γιατί ε, έχουμε εισαγάγει τέτοια οδηγία όπω και άλλοι. Τι θα κάνει η Κομισιόν τόσο ώστε να εξασφαλίσει ότι τέτοιου τύπου νομοθεσία ανακαλείται το συντομότερο δυνατόν στα κράτη μα. Και έπειτα υπάρχει και η συμφωνία SWIFT, που είναι βασίζεται στι ίδιε αρχέ όπου γίνεται μαζική ε, διατήρηση δεδομένων, χίδιν, για ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα, καμία αξιόπινη πράξη. Ε, πολλές φορές σας ζητήσαμε, κυρία Μάστον, να σταματήσετε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τι θα κάνετε για όλα αυτά. Τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στην κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπήρξε μια σύγχυση γι' αυτό ήρθα καθυστερημένα. Θα ήθελα να χαιρετήσω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει προφανώς ε, συνέπειες όχι μόνο για την οδηγία αλλά και για την εθνική νομοθεσία που προήλθε από την οδηγία. Και εδώ πρέπει η Κομισιόν να παρέμβει ώστε να εξασφαλίσει ότι τα εθνικά κοινοβούλια, τα εθνικά μάλλον δικαστήρια, θα σεβαστούν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτή η απόφαση έχει σημασία για τι διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων και είναι απαραίτητο οι διαπραγματεύσει αυτέ να εξασφαλίσουν το δικαίωμα νομικής προσφυγής, δικαστικής προσφυγής, συγγνώμη, σε, δικαστικό, σε διοικητικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως ακριβώς γίνεται και για τους Αμερικανούς πολίτες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος τώρα, Μάστρομ, θα κάνει τις ε, καταληκτικές της ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτέ για αυτή τη συζήτηση. Όπως είπα και στην αρχή, η Κομισιόν καλωσορίζει την απόφαση του δικαστηρίου Ούτω ή άλλω και πριν από κάνα δύο χρόνια κάναμε τη δική μα αξιολόγηση και είχαμε πει παρόμοια πράγματα. Αξιολογούμε τώρα τι επιπτώσει απόφαση. Χρειάζεται χρόνο. Πρέπει να αξιολογήσουμε ε, προσεκτικά με του εμπειρογνώμονέ μα τι επιπτώσει αυτέ. Κάποια πράγματα όμω είναι σαφή ήδη. Όπω είπατε, καταρχήν, η δήλωση για την ακυρότητα ε, αρχίζει να ισχύει πάρα αυτά. Την ε, ημέρα δηλαδή, από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία. Δηλαδή ουσιαστικά φτάσαμε στην κατάσταση πρώτου 2006 πριν υιοθετηθεί η οδηγία. Γι' αυτό η Κομισιόν θα κάνει ό,τι πρέπει για να σταματήσει η δίωξη της Γερμανίας και τα πρόστιμα που κατέβαλε η Σουηδία θα επιστραφούν. Επίσης, από την απόφαση προκύπτει ότι η Εθνική Νομοθεσία των Κρατών Μελών είναι άσχετη, όχι τουλάχιστον άμεσα σχετική με την απόφαση. Κάθε κρατό μέλο θα πρέπει να αξιολογήσει μήπω πρέπει να αλλάξει την εθνική νομοθεσία. Και οι, Ευρωπα... οι εθνικέ αρχέ θα αποφασίσουν εάν η δική του νομοθεσία ε, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ακούστηκαν κάποιε ερωτήσει τώρα για το PNR και τη συμφωνία TTIP με τι ΗΠΑ. Αξιολογούμε πολύ προσεκτικά και επανεξιολογούμε αυτές τις συμφωνίες. Από ό,τι Φαίνεται όμως ε, έχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες οι συμφωνίες αυτές και επανεξετάζονται τακτικά από δικές ομάδες και νομίζουμε ότι έχει καμία σχέση οι, συμφωνίε οι συμφωνίες αυτές με την απόφαση του δικαστηρίου θα επανέλθουμε. Σε ό,τι αφορά την οδηγία, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το PNR που πρότεινε η Κομισιόν και έχουμε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Ολομέλεια. Αυτά τα δύο θέματα δεν είναι συγκρίσιμα. Η προτινόμενη οδηγία για το PNR αφορά όλα τα, ε, διασκεδάζει όλες αυτές τις ανησυχίες και όλα τα προβλήματα που θέτει η απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί ε, περιορίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα και η χρήση τους. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι ειδικοί. Η χρήση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να καταπολεμήσουμε σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία και οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων απαγορεύεται. Επίση, η πρόταση έχει ασφαλιστικέ δικλείδε αποτελεσματικέ για να προστατεύονται τα δεδομένα. Όπω σα είπα, θα συνεργαστούμε μαζί σας, με το επόμενο κοινοβούλιο φυσικά, για την ε, πρόταση μιας οδηγία, της οδηγίας PNR και θα αξιολογήσουμε μαζί εάν ε, η σαφή οριοθέτηση ε, είναι επαρκή οριοθέτηση είναι υπόψη μα όσου θα είπε ή πρέπει να υιοθετηθούν και άλλα μέτρα. Θα λάβουμε υπόψη μας τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα εμπνευστούμε από αυτά. Τώρα, είναι πολύ νωρίς να σκεφτούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά τα πράγματα, κύριε Βέμπερ. Εάν γίνει μία πρόταση, αν προτείνουμε κάτι νέο από πλευρά Κομισιόν, εάν το υπογραμμίζω, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη φυσικά τι επιπτώσει τη απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά και τα θέματα προστασία των δεδομένων που έχετε πει πολλέ φορέ, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο αυτό. Ε, πριν από καμιά ε, δύο εβδομάδες συζητήσαμε το πρόγραμμα μετά τη Στοκχόλμη και το θέμα της ασφαλού Ευρώπης. Και στην, στο έγγραφο που σα δώσαμε είχαμε πει ότι θα αναθεωρήσουμε την απόφαση αυτή για την, την οδηγία συγγνώμη, για την διατήρηση των δεδομένων, μάλιστα πριν την απόφαση του δικαστηρίου. Και αν χρειαστεί, θα κάνουμε μια πρόταση νέου τύπου, λαμβάνοντα υπόψη τα όσα είπε το δικαστήριο. Όλα αυτά θα ακολουθήσουν την κλασική νομοθετική διαδικασία, με πλήρη δηλαδή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ νωρίς για να τα προδικάσουμε. Θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό το θέμα όταν θα έχουμε αναλύσει όλες τις νομικές επιπτώσεις της απόφασης του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Κλείνει η συζήτηση. Επόμενο σημείο τη μέσα διάταξη είναι δήλωση από την Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή και είπα την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφαλεία με θέμα θρησκευτικέ ελευθερίε ε, και πολιτιστική διαφορετικότητα. Πρώτο ομιλητή ο κύριο Κούρκουλα, εκ